η ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Όχι. Αποτείουμε φόρο τιμής ε, στα πάνω από 5.000 θύματα που είχαμε στην Ευρώπη και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας για τους ε, πάρα πολλούς ανθρώπους που υπήρξαν θύματα ή ε, τραυματίστηκαν και υπέστησαν τις ε, ζημίες της τρομοκρατίας. Τα όσα είχαμε στη Μαδρίτη πριν από έξι χρόνια, στις 11 Μαρτίου του 2004, τα οποία προκάλεσαν το θάνατο 191 ατόμων από 17 χώρες και οι βόμβες οι οποίες εξερέγησαν στο Λονδίνο στις 7 Ιουλίου του 2005 θεωρούνται από τις ε, χειρότερες τρομοκρατικές ε, πράξεις που έχουν γίνει ποτέ σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η τρομοκρατία είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας. Είναι μια απόπειρα κατά του ιστού της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρώπη θα είναι πάντα ενωμένη στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας ε, διαχωρισμός θρησκευτικός ή πολιτικός. Ποτέ δεν υπάρχει αιτιολόγηση για την τρομοκρατία με κανένα τρόπο και με κανένα λόγο. Αυτή η Ευρωπαϊκή ημέρα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να αποδείξουμε ότι κανένας τρομοκράτης και καμία τρομοκρατική πράξη δεν θα μπορέσουν ποτέ να καταστρέψουν και να ε, διακυβεύσουν την πίστη μας στις βασικές αρχές, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα θεμελιώδη δικαιώματα και στη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Cari colleghi, nel corso della sua riunione... Αγαπητοί συναδελφοί, στα σημερινή της συνεδρίαση η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε βάσει του άρθρου 134 παράγραφος 3 του κανονισμού μας να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα των ε, Ολομελιών και να συγκαλέσει συνεδρίαση για την ε, Τετάρτη 7 Απριλίου 2010 από τις 2.30 έως τις 4.30 το απόγευμα. Η ημερήσια διάταξη της ε, Συνόδου θα περιλαμβάνει μία έκθεση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης και 26ης Μαρτίου 2010.